Η σύνοδος θα συνεχιστεί αύριο από τις 8.30 ε, το πρωί. Η μερίστη διάταξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να ευχαριστήσω την